Τελειώσαμε, συνάδελφοι, την σημερινή συνεδρίαση. Αύριο θα έχουμε τη νέα συνεδρίαση, 13 του μηνός, 9 με 1, ως συνήθως, 3 με 7 και 9 με 12 τη νύχτα. η σε διάταξη είναι στο σχετικό έγγραφο και μπορείτε να δείτε την ημερήσια διάταξη και στο ίντερνετ. Καλή σας νύχτα και ευχαριστώ για την προσοχή σας.